διαφορετική αντιμετώπιση των μεν και των δε, αλλά υπάρχει και μία θέση της πλειοψηφίας, η οποία θέση της πλειοψηφίας είναι περαιτέρω εκτίμηση και αξιολόγηση αυτών των αριθμών. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Τουρίπελη. Έτσι ολοκληρώνεται η κοινή συζήτηση για το προπολογισμό. Ευχαριστώ όλου για τις παρεμβάσεις τους. Περαιούτη η συζήτηση. Η ψηφοφορία τη έκθεση Μάνκα θα γίνει αύριο και η έκθεση τη κυρίας Τρίπελ σήμερα το μεσημέρι. Προχωρούμε τώρα στην ακόλουθη συζήτηση με βάση την μερίση διάταξη κοινή συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν με την έκθεση Τάβαρες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων για την περίοδο 2008 έως 2013 και την έκθεση Σεϊνό, Κοέλιο, συγγνώμη, για την μετάβαση από το σύστημα πληροφοριών Σέγγεν 1 στο SIS 2 καθώς και τη μετάβαση από το σύστημα Σέγγεν 1 στο σύστημα πληροφοριών Σέγγεν 2, επιπλέον δε και την έκθεση Τάβαρης για τη δημιουργία ενός κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος επανεγκατάστασης. Ξεκινούμε με την συζήτηση για το σύστημα Σέγγεν και Δίνω το λόγο στον κύριο Κοέλιο. Κάπως ε, έφαγα το όνομά σας, συγγνώμη, ο οποίος είναι συνεισηγητής για τέσσερα λεπτά. Παρακαλώ. Πολύ καλά το είπατε το όνομά μου, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ξεκινήσω υπενθυμίζοντας ότι το Κοινοβούλιο ήδη αναφέρθηκε στι καθυστερήσει στο πρόγραμμα αυτά, αυτό. Το 2009 εγκρίναμε ένα ψήφισμα για το ε, σύστημα πληροφοριών Schengen 2 και το, σύστημα, και το VIS, το σύστημα πληροφοριών για τις θεωρήσεις. Και είχαμε εκφράσει την ανησυχία μας για την καθυστέρηση που διαπιστώνεται στην έναρξη δραστηριοτήτων και στην καθυστέρηση στις τεχνικές λεπτομέρειες και ζητούσαμε να υπάρχει διαφάνεια σε ό,τι αφορά την υλοποίηση του SIS 2. Το 2007 είχαν γίνει αυτά. Τώρα είμαστε στο 2010 και κανείς δεν εγγυάται πότε θα ολοκληρωθεί η διαδικασία. Σε σχέση με το πακέτο που εξετάζουμε, δημιουργούνται τέσσερις βασικές ερωτήσεις. Πότε θα ολοκληρωθεί η μεταφορά αυτή, ε, η μετάβαση αυτή. Η θέση σε ισχύ θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον διαπιστωθεί ότι το σύστημα τηρεί όλες τις προϋποθέσεις του νομικού εργαλείου. Όταν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα μπορέσει να γίνει η μετάβαση από το SIS-1 στο SIS-2. Έχουν τελειώσει οι δοκιμές αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν προβλήματα και δυσκολίες ε, όπως διαπιστώθηκαν από τις δοκιμές. Για το λόγο αυτό το Συμβούλιο αποφάσισε νέες ε, δοκιμές του 2009. Το πρώτο τεστ έγινε τον Ιανουάριο γιατί δεν είχαν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις. Τον Ιανουάριο του 2010 εννοώ. Στις δοκιμές αυτές διαπιστώθηκε ότι το σύστημα δεν είναι σταθερό. Επανε... Επαναλήφθηκαν οι δοκιμές από τις 2 στις 5 Μαρτίου. Η αξιολόγηση των ε, δοκιμών έγιναν τον Απρίλιο. Παρότι οι συνθήκες των δοκιμών, ε, οι προϋποθέσεις των δοκιμών δεν τηρήθηκαν πλήρως και παρότι ε, οι χρονικές ε, προθεσμίες απάντηση που απαιτήθηκαν δεν τηρήθηκαν επίση. Τα κράτη-μέλη κατέληξαν παρόλα αυτά στο συμπέρασμα ότι και με τα προβλήματα αυτά οι δοκιμές είχαν αποβεί ε, επιτυχής. Επίσης θεωρήθηκε αναγκαίο οι υπόλοιπε προποθέσει να τηρηθούν πριν το ξεκίνημα των νέων ε, της νέας διαδικασίας. Θα πρέπει το SIS2 να λειτουργεί σωστά και θα πρέπει να είναι επιτυχής και η δοκιμή που προβλέπει το άρθρο 55 εξασφαλίζοντας την ε, ακαιρεότητα και την ασφάλεια του δικτύου. Τώρα, γιατί βιαζόμαστε για την έγκριση των ε, πρωτοβουλειών αυτών παρότι οι προϋποθέσεις για τη μετάβαση δεν είναι πλήρως ολοκληρωμένες. Η εντολή που είχε αναλάβει η Κομισιόν για το SIS-2 λήγει φέτος τον Ιούνιο. Συνεπώς θα πρέπει να αλλάξουν οι ρήτρε ακύρωσης που είχαν προβλεφθεί το 2008 για να μην ε, εκπνεύσει η εντολή προς την Επιτροπή. Άλλη ερώτηση. Τι αλλάζει η πρόταση αυτή. Καταρχάς υπάρχει μια ρήτρα ε, που δεν είχε προτείνει η Επιτροπή. Εμείς θεωρούμε αυτό να είναι τον Δεκέμβριο του 2011. Είναι αναγκαίο και λόγω των καθυστερήσεων. Θα πρέπει η νομική βάση να επιτρέπει την βελτίωση, τη χρήση της καλύτερης δυνατής υφιστάμενης ε, τεχνολογίας και με ένα αποδεκτό χρονοδιάγραμμα ταυτόχρονα. Θα πρέπει να υπάρχει μια συνολική διαχείριση του συστήματος. Είμαι πεπισμένος ότι αν είχε υπάρξει ένα όργανο ε, διαχείριση του συστήματος εξ αρχής είχαμε προχωρήσει καλύτερα. Πιστεύω ότι η μετάβαση αυτή πρέπει να υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο. Το Κοινοβούλιο δεν είναι υπεύθυνο μόνο για τη νομική βάση. Εξασφαλίζει ταυτόχρονα και την έγκριση των δράσεων που έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον συνάδελφο κύριο Άλβαρο ζητήσαμε η κυρία Λάτφορντ και η κυρία Μάγερ όλοι μαζί να μπουν τα ποσά στο αποθεματικό και να υπάρξει αξιολόγηση από το ελεκτικό συνέδριο. Ο κύριος Σταβάρης είχε κάποια προβλήματα μετακίνησης λόγω κάποιου ηφαιστείου αλλά και δεν είναι εδώ. Μόλις έρθει ωστόσο θα του δώσω το λόγο. Θα δώσω κατευθείαν το λόγο στον κύριο Άλβαρο τώρα από την Επιτροπή Προπολογισμών για ένα λεπτό. Το SIS 2, το σύστημα πληροφοριών Schengen δεύτερης γενιάς, είναι μια μακρά ιστορία δοκιμών, αποτυχιών και ε, ε, ε, δαπανήθηκαν δεν 90 εκατομμύρια ευρώ και πρέπει να πω ότι παρακολούθησα κάθε βήμα που έκανε ο συνάδελφος κύριος ε, Κουέλιο ε, και συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Αλλά όπως όλα τα πράγματα στη ζωή πρέπει να παραδεχθούμε ότι τα πράγματα δεν ε, λειτουργούν έτσι όπως θέλουμε κάποια στιγμή και πρέπει να αναζητήσουμε νέες εναλλακτικέ. Ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε έτοιμοι να εγκαταλείψουμε το project Από την άλλη, ο Επίτροπος μας είπε ότι θέλει να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Από την άλλη, όμως, θα πρέπει να υπάρχει καλύτερος έλεγχος των χρημάτων που δαπανώνται. Αυτή τη στιγμή ε, καταρτίζεται ένα δεύτερο πρόγραμμα το οποίο ξέρουμε ότι δεν θα λειτουργήσει. Για ποιο λόγο το κάνουμε. Και τώρα, ε, απουσία της κυρίας, ε, του κυρίου Ταβάρες, δίνω τον λόγο στην Επίτροπο κυρία Μάστρο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ε, αρχίζω με το δεύτερο και θα επανέλθουμε στην έκθεση Ταβάρες. Ε, πώς θα γίνει. Ωραία. Αξιότιμα μέλη αξιότιμοι κύριοι Κουέλιο και Αρβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ για τις παρεμβάσεις σας και για τον επικοδομητικό τρόπο με τον οποίο συνεργαστήκατε σε αυτό το πάρα πολύ σύνθετο φάκελο που κληρονόμησα. Πράγματι πολύπλοκο και σύνθετο. Ωστόσο είμαι αποφασισμένη να συνεργαστώ μαζί σας για να προχωρήσουμε με διαφανή τρόπο και να ολοκληρώσουμε το έργο. Πράγματι η συζήτηση είναι πολύ έγκαιρη. Επιβεβαίωσε το Συμβούλιο ότι το, η πρώτη δοκιμή ήταν επιτυχής και θα συνεχίσει συζητήσουμε επί τη βάση των υπαρχόντων τεχνικών λύσεων. Η πρόταση λοιπόν που έχετε ενώπιόν σας περιέχει τρία βασικά στοιχεία στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Κουέλιο και τούτο θα μεταβάλει την εξέλιξη του προγράμματος. Πρώτον, όπως είπε ο κύριος Κουέλιο, η προθεσμία 30 Ιουνίου δεν είναι ρεαλιστική και συνεφώς αλλάζει. Τούτο θα επιτρέψει έργο να προσαρμοστεί στις τεχνικές προδιαγραφές τα οποία θα επαναπροσδιοριστούν σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμενες των χωρών μελών και θα είναι στη διάθεση του Συμβουλίου 3 και 4 Συμβουλίου. Ο εισηγητής αναφέρει συγκεκριμένη προθεσμία. Λυπούμε που η Κομισιόν αυτή τη στιγμή δεν είναι σε θέση να δεχτεί την πρόταση αυτή. Οι εμπειρογνώμενες της Κομισιόν μαζί με τις χώρες μέλη αυτή τη στιγμή εξετάζουν την οριστικοποίηση των προδιαγραφών ε, στο πλαίσιο ενός νέου χρονοδιαγράμματος. Από τη στιγμή που τούτο θα συμβεί θα καθοριστεί αυτό το πρόγραμμα και θα υποβληθεί στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων σε δύο εβδομάδες. Το, η ομάδα, μάλλον το Συμβούλιο, το Συμβούλιο δύο. είναι ένα διοικητικό συμβούλιο συνολικού προγράμματο, ε, το οποίο συνεχίζει το έργο του, είναι μια ομάδα εργασία, για να εξετάσει τι διαδικασίες και τις προϋποθέσεις. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά τεχνικό σώμα. Δεν χρειάζεται να ανοίξει σε άλλα στελέχη ή βουλευτέ. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε με διαφανή τρόπο σε συνεργασία με το Κοινοβούλιο και να κάνουμε σαφή διάκριση μεταξύ τη τεχνικής δουλειά και τη πολιτική διαφάνεια. Με το πνεύμα αυτό η Κομισιόν είναι έτοιμη να προσφέρει ε, ε, πλήρη τεχνική αρρωγή στα μέλη του Κοινοβουλίου και βάσει των ε, συστάσεων αυτού του Τεχνικού Συμβουλίου όπως προτείνει ο κύριος Κουέλιο. Η απαραίτητη νομική ευελιξία που απαιτείται για ένα εναλλακτικό σενάριο θα προβλεφθεί και νομίζω ότι τούτο θα είναι μια ορθολογική επιλογή. Ω προ τι δημοσιονομικέ ε, πτυχέ, για συνέχιση του έργου, η Κομισιόν συμμερίζεται την άποψη του εισηγητή ότι θα πρέπει να κάνουμε βέλτιστη χρήση των χρημάτων των φορολογουμένων. Από την άλλη διατηρείται το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ορίζει ε, το ύψος ε, των ποσών που θα τεθούν στα αποθεματικά του προϋπολισμού 2011. Τώρα, σχετικά με την ε, εφαρμογή του προϋπολογισμού θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Άλβαρο να προβλέψει μια λογική διαδικασία απεμπλοκής όταν τα κονδύλια θα είναι απαραίτητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κουέλιο και τον εισηγητή στην Επιτροπή, τον κύριο Άλβαρο, για την εξαιρετική συνεργασία επ' αυτού του φακέλου. Επιτρέψατε μου τώρα, κυρία Πρόεδρε, να πω ακόμα δύο λόγια. Λυπάμαι που ο κύριος Αλβάρε δεν είναι παρόν ε, για να συζητήσουμε μαζί του σε αυτό το ε, πολύ σοβαρό θέμα. Όπω γνωρίζετε, μεγάλο αριθμό μεταναστών έρχονται σε... μεγάλο αριθμό προσφύγων ε, φιλοξενούνται σε διάφορες ε, χώρες, σε ε, άσχημη κατάσταση. Δεν μπορούν να επιστρέψουν στις χώρες προέλευσης, ούτε μπορούν να ενταχθούν στις χώρες πρώτου ασύλου, διότι και αυτές οι ίδιες χώρες είναι θύματα φτώχειας. Και άρα λοιπόν η επανεγκατάστασή του είναι η μόνη λύση σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση και τούτο θα ήταν μια πολύ συγκεκριμένη ε, ένδειξη αλληλεγγύη σε αυτές τι χώρες πρώτου ασύλου και με αυτόν τον τρόπο θα προσφέρουμε προστασία σε, στους πιο ευάλωτους ε, από αυτούς τους πρόσφυγες. Αυτή τη στιγμή ωστόσο δεν υπάρχει διαρθρωτικό συντονισμός μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Κομισιόν θεωρεί ότι μπορούμε να διαδραματίσουμε μεγαλύτερο ε, και καλύτερο ρόλο ενισχύοντας τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκοσμίω και επιδεικνύοντας και την απαραίτητη αλληλεγγύη. Η πρόταση που υποβλήθηκε το Σεπτέμβριο του 2009 έχει ως στόχο τη βελτίωση της κατάστασης. Ικανοποιούμαστε από τη την θετική ανταπόκριση που επέδειξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στην πρόταση αυτή. Και ευχαριστώ τον κύριο Ταβάρες για, την, ε, για το έργο του και την ισχυρή πολιτική συνένεση μεταξύ των πολιτικών ομάδων στο θέμα αυτό. Η ιδέα στην πρόταση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με την ύπατη αρμοστία του ΓΕ για τους ε, ε, πρόσφυγες να συνεργαστεί σε μια στρατηγική ε, διάστασης ε, ε, λύση σε αιτήσια βάση. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αμβλύνουμε την κατάσταση σε κάποιες από τις περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις. Θα, η τελική πρόταση προβλέπει η τελική επιλογή, ο αριθμός των προσφύγων να καθοριστεί ανάλογα με τη βάση και τη γνώση που υπάρχει σε κάθε χώρα. Έτσι λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να αντιδρά καλύτερα τις αυξανόμενες προκλήσεις ε, όσον αφορά τους πρόσφυγες και θα καταστήσει πιο αποτελεσματικές, Προεποτελεσματική τη λειτουργία ε, του Ειδικού Ταμείου για τους ε, πρόσφυγες ώστε να βοηθηθούν οι χώρες που δέχονται τους πρόσφυγες. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν και η κοινωνία θα ανταποκριθεί καλύτερα. Συμφωνώ λοιπόν με την, με την πρόταση του συγητή για ένα ειδικό γραφείο στην Μάλτα. Από το 2007 πέντε χώρες μέλη μαζί με εκείνες που ήδη είχαν προγράμματα αποφάσισαν να ε, εφαρμόσουν προγράμματα, εθνικά προγράμματα επανεγκατάστασης και έχουν δεχθεί πρόσφυγες από το Ιράκ σε ανταπόκριση της δέσμευσης που ελήφθη το 2008. Είναι κρίσιμη σημασία να ανταποκριθούμε σε αυτή την ε, κρίσιμη στιγμή. Λυπούμαστε ωστόσο ότι υπάρχουν αποκλήσεις ως προς τα διαδικαστικά και χρειάζεται μια ταχεία υιοθέτηση της πρότασης αυτής που έχει τεράστια πολιτική σημασία. Η απόφαση της Κομισιόν να θεσπίσει ετήσιες προτεραιότητες για την επανεγκατάσταση είναι ε, πρακτικού χαρακτήρα, όπως επίσης και ε, σε σχέση με τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων. Εμάς μας ενδιαφέρει η διαδικασία αυτή μας ενδιαφέρει το γεγονός ότι καθυστερεί η διαδικασία και η διάθεση των κονδυλίων καθυστερεί. Άρα λοιπόν θέλουμε να έχουμε μια κοινή προσέγγιση, μια επανεξέταση της προσέγγισης θα γίνει, είναι φιλόδοξα τα σχέδια ε, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Θα δώσω τώρα το λόγο στους συζητητές εξ ονόματος των ομάδων και αρχίζω με τον κύριο Παπα-Νικολάου για δύο λεπτά εξ ονόματος του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για την ενημέρωσή σας. Παρότι ο κύριος Σταβάρες δεν είναι μαζί μας, ε, θέλω να τον ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι σήμερα και πράγματι ε, να εκφράσω και εγώ την δική μας θετική τοποθέτηση από την πλευρά της δικής μας πολιτικής ομάδας ε, σε σχέση με το πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Αναφερόμαστε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σε ένα ενιαίο χώρο για το άσυλο και σε μια ολοκληρωμένη πολιτική διαχείρισης προσφύγων την οποία πρέπει να έχουμε. Και βεβαίως το χρηματοδοτικό εργαλείο για να στηρίξει αυτή την προσπάθεια είναι το ευρωπαϊκό ταμείο για τους πρόσφυγες το οποίο μέχρι σήμερα η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε εξαντλήσει επαρκώς και υπάρχουν περιθώρια για να κάνουμε ακόμη πιο σημαντικά πράγματα. η ευρωπαϊκή ανταπόκριση στις παγκόσμιες ανάγκες για την επανεγκατάσταση μέχρι σήμερα είναι επαρκή. υπενθυμίζω ότι η συμμετοχή των κρατών μελών είναι σε εθελοντική βάση και μέχρι σήμερα μαζί με τις δύο χώρες που ad hoc έλαβαν μέρος στην επανεγκατάσταση έχουμε μόνο δώδεκα από τα 27 κράτη μέλη να συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια με αριθμού οι οποίοι δεν είναι ιδιαίτερα καλοί μέχρι σήμερα έξι έξι πρόσφυγες το 2009 έφτασαν στην Ευρώπη με το πρόγραμμα επανεγκατάστασης που αντιπροσωπεύουν μόνο το 8,2%. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε σίγουρα καλύτερο συντονισμό και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε μέσα από αυτήν την έκθεση και τη διαβούλευση που είχαμε ήταν να δώσουμε κίνητρα, να εξηγήσουμε στα κράτη-μέλη ότι έχουμε κάθε λόγο να προχωρήσουμε στην εφαρμογή και υιοθέτηση αυτού του προγράμματος. Βεβαίω, η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η έμπρακτη αλληλεγγύη μα προ τι τρίτε χώρε είναι ε, στόχευση ε, πρώτης προτεραιότητας πρέπει όμως να γίνει αντιληπτό ότι ένας ακόμη λόγος που όλα τα κράτη μέλη έχουν λόγους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό είναι γιατί μέσα από αυτό το πρόγραμμα μπορούμε να δώσουμε σε όλους εκείνους που έχουν ανάγκη το μήνυμα ότι έχουν κάθε λόγο να επιλέγουν νόμιμες οδούς για να προσπαθούν να φτάσουν ε, την ευρώπη το ευρωπαϊκό έδαφος για μια καλύτερη τύχη. θέλω να πω και με συγχωρείτε κυρία πρόεδρε ότι η παράνομη μετανάστευση έμεσα μπορεί να αντιμετωπιστεί και μέσα από τα προγράμματα επανεγκατάστασης με την έννοια ότι ε, με αυτά τα προγράμματα ο πρόσφυγας δεν θα επιλέξει παράνομους οδούς αλλά θα περιμένει να ενταχθεί στα προγράμματα αυτά. τέλος και κλείνω ε, κάναμε μια τροπολογία η οποία δεν προχώρησε σε σχέση με την εσωτερική επανεγκατάσταση προσφύγων. κάποια στιγμή κυρία επίτροπε αναμένουμε πρωτοβουλία της επιτροπής σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Είναι κάποιες χώρες και είναι πολύ σημαντικό από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων να προχωρήσουμε στο Καταλάβατε νομίζω. Ευχαριστώ. Και δίνω το λόγο στον κύριο Μασί Δάλγο. Ενάμιση λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ την κυρία Μάλσον για την παρουσία της εδώ. Θέλω να συμφωνήσω με την έκθεση και με το πνεύμα της δουλειάς του κυρίου Ταβάρες. Η δουλειά του με τις ΜΚΟ, με την ΑΡΜΟΣΤΙΑ, με την συγκριτική προσέγγιση της νομοθεσίας των χωρών εκτός της Ένωσης είναι πολύ σημαντική. Είναι σημαντικές αυτές οι βασικές ε, ε, προϋποθέσεις και θέλω ε, ήμουν ε, σε ένα δήμο παλιά και θα ήθελα να μετάσχουν στη δραστηριότητα αυτό όλοι οι δήμοι της Ευρώπης γιατί βιώνουμε μια κρίση η πιο βαθιά ωστόσο κρίση στην ιστορία του ασύλου και των προσφύγων. Υπήρχε, υπάρχει μια κτίση συνολικής αμνησίας. Ξεχάσαμε στην Ευρώπη, στις πλούσιες χώρες, το ότι οι πόλεμοι που δημιουργούν τους πρόσφυγες είναι δική μας ευθύνη ευθύνη των χωρών και των κρατών μας και των κυβερνοϊσών μας. Αυτή την συλλογική αμνησία πρέπει να την ε, ξεπεράσουμε. Συμφωνώ με την κυρία Μάλστρομ. Πρέπει η Επιτροπή ε, να, να δουλέψουμε στον τομέα αυτό. Υπήρξε μια πίσκεψη επίσκεψη βουλευτών του Κοινοβουλίου στους Παλαιστίνιους στα, σε στρατόπεδο όπου κατοικούν Παλαιστίνοι του Ιράκ. Ε, πρέπει, επαναλαμβάνω πρόεδρε, να ξεπεραστούν οι διαφορές μεταξύ Κοινοβουλίου, ήσασταν βουλευτής εσείς και Επιτροπής για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Δεν θα ήθελα η έκθεση σήμερα να ε, είναι μια ε, διαδικασία που τελικά θα μπλοκαριστεί γιατί το Κοινοβούλιο δεν συμφωνεί με τη δική σας αντίληψη για τις κατεξουσιοδότηση πράξεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Χίος για τους φιλελεύθερους. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Πίτροπε. Πιστεύω ότι όλα όσα άκουσα δείχνουν ότι θα πρέπει πραγματικά να συμμετάσχουν όλο και περισσότερα κράτη στην επίληψη αυτών των θεμάτων. Θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής σε ένα σύστημα. Όλοι όσοι μέχρι τώρα συμμετείχαν έχουν υπογραμμίσει αυτά τα θετικά. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά τα άτομα τα οποία φτάνουν στην Ευρώπη, τα οποία ζουν στα στρατόπεδα προσφύγων, τα οποία χρειάζονται την βοήθεια και την υποστήριξή μας, είναι γυναίκες, είναι παιδιά, είναι ηλικιωμένοι, είναι άρρωστοι και θα πρέπει να δούμε τι ποσά έχουμε στη διάθεσή μας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει εδώ επίξης να παίξουν το ρόλο τους. Δηλαδή τα κονδύλια αυτά να μην εξαφανίζονται σε άλλες δραστηριότητες, αλλά πραγματικά να χρησιμοποιηθούν για όλη αυτή την προσπάθεια και τη δημιουργία υποδομών, για τη δημιουργία σχολείων, βρεφή. Φωνηπιακών σταθμών, νοσοκομείων, περίθαλψης. Τα κράτη προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το θέμα αυτό με βραχυπρόθεσμη σκοπιά, να το αρνηθούν, να το καλύψουν. Εμείς όμως, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει πραγματικά να δημιουργήσουμε αυτές τις δομές της ενσωμάτωσης όλες αυτές τις απαραίτητες υποδομές οι οποίες θα οδηγήσουν όλους αυτούς τους ανθρώπους να ενσωματωθούν στις κοινωνικές μας. Και θα πρέπει να εξηγήσουμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι τα άτομα αυτά τα οποία θέλουν να ξεκινήσουν μια καινούρια ζωή να το κάνουν με εύκολο τρόπο σε κράτη στα οποία προβλέπεται η περίθαλψή τους, η ενσωμάτωσή τους και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με νέα προγράμματα και με μια νέα αντιμετώπιση. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα στηρίξουμε αυτή την πολιτική της ενσωμάτωσης. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Έχω ένα τεχνικό πρόβλημα εδώ, γι' αυτό και δεν μπόρεσα να σας διακόψω, αλλά ευτυχώς καταλάβατε το μήνυμά μας. Η κυρία Φλότ, εξ ονόματος των Πρασίνων, για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ο κύριος Ταβάρες άργησε, αλλά επιτέλους ήρθε. Νομίζω ότι η εργασία του για να βρεθεί μια συνένεση, μια συμφωνία όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους πρόσφυγες, όσον αφορά την βοήθεια που θα πρέπει να προσφέρουμε στους πρόσφυγες, είναι μια εξαιρετική προσπάθεια και η Επίτροπος την στηρίζει. Θα ήθελα να αναφέρω κάποιους αριθμούς. Εάν δαπανίσουμε κάτι το οποίο βεβαίως και δεν το επιθυμώ, γιατί αυτά τα χρήματα θα βγουν από κάπου αλλού, εάν δαπανηθούν όλα τα ποσά που διατίθεται, θα μπορέσουμε να στηρίξουμε και να ενσωματώσουμε περίπου 20.000 πρόσφυγες μόνο. Τίποτα δηλαδή σε σχέση με τους 400.000 πρόσφυγες που περιμένουν τη στήριξή μας, άτομα τα οποία είναι ευάλωτα, τα οποία δεν μπορούν να γυρίσουν στις χώρες από τις οποίες προέρχονται. Δεν έχουν τη δυνατότητα. Στην Γαλλία, στη χώρα μου, έχουμε μία εμπειρία όσον αφορά την ενσωμάτωση κάποιων ελάχιστων προσφύγων γιατί όπως ξέρετε οι επιτυχημένες προσπάθειες στη Γαλλία είναι ελάχιστες και κρύβουν ένα μεγάλο αριθμό απάνθρωπων πρακτικών. Δεν ξέρω να ξέρετε ότι η χώρα μου μόλις καταδικάστηκε για βασανισμούς και απάνθρωπη αντιμετώπιση προσφύγων. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Φλότρ. Η κυρία Βράζια έχει το λόγο, εξ ονόματος των αριστερών, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να παρέμβω σχετικά με το σύστημα πληροφοριών Schengen. Θα πρέπει σήμερα να εξετάσουμε το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μας επιτρέψει να μετατρέψουμε το σύστημα προς την κατεύθυνση του ΣΥΣ 2. Το ελάχιστο που μπορούμε να πούμε, κυρία Επίτροπε, ε, είναι ότι οι δοκιμές δεν έχουν ολοκληρωθεί επί του θέματος. Ωστόσο, ε, θα πρέπει να δούμε τη θέση των τριών χωρών, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία. Στο πλαίσιο της ε, ομάδας ΓΚΟΕ γνωρίζετε ότι έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Επίμονες επιφυλάξεις μάλιστα όσον αφορά το ζήτημα της εγγραφής και τούτο συνδέεται άμεσα και με την προστασία των δεδομένων. Ασφαλώς πρέπει να είμαστε ε, ρεαλιστές ε, και να δούμε τους πραγματικούς κινδύνους ε, που υπάρχουν όσον αφορά στα ζητήματα ασφάλειας και να ακούσουμε αυτά τα οποία μας λένε οι ειδικοί. Θα πρέπει να λάβουμε μέτρα για την προστασία των δεδομένων για όλους τους πολίτες όποιοι και αν είναι αυτοί. Και θα πρέπει να έχουμε ένα ελάχιστο δέσμευση ε, για δέσμευση όσον αφορά τον κίνδυνο της διασύνδεσης των κατολόγων. Ε, άρα λοιπόν υπό την παρούσα ε, κατάσταση η ομάδα μας δεν είναι σύμφωνη με μια τέτοια μετάβαση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπάτον για 1,5 λεπτό. Η Βρετανία, κυρία ε, Πρόεδρε, δεν είναι εγγεγραμμένη στο Σέγγεν και συνεπώς η πρόταση δεν θα εφαρμοστεί στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η προηγούμενη κυβέρνηση των εργατικών δεν εντάχθηκε και η νέα κυβέρνηση συμμαχίας δεν πιστεύω ότι είναι υπέρ της άποψης αυτής. Για φανταστείτε όταν θα ενταχθεί η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναμένουμε όχι μόνο τα 72 εκατομμύρια των Τούρκων που θα έχουν αυτόματη είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ηνωμένο Βασίλειο αλλά επίσης και ε, μια πλημμυρίδα ε, προσφύγων από χώρες όπως το Ιράκ και άλλες χώρες προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Βρετανία αντιτίθεται σε ένα τέτοιο ε, σχέδιο. Ωστόσο, το ίμιση του ε, το ίμιση του συντηρητικού κόμματος ε, δηλώνουν σκεπτικιστές, ε, ό,τι σημαίνει αυτό, και το άλλο είναι ευρωφοβική. Εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια πλήρης αναθεώρηση της συνθήκης της Λισαβόνας. Ο κύριος Κάμερον μπορεί να επιλέξει είτε να μην επικυρώσει είτε να ζητήσει τα απαραίτητε εγγυήσεις με ένα δημοψήφισμα που θα οργανώσει μεταξύ του Βρετανικού λαού. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής, εξονόμενος των... της Επιτροπής των Ελευθεριών, έχει το λόγο, ο κύριος Τάβαρες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν, θα ήθελα να πω ότι παντού στον κόσμο υπάρχουν πρόσφυγες οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις χώρες τους και δεν μπορούν και να εγκατασταθούν και να εργαστούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για 200.000 πρόσφυγες οι οποίοι επιθυμούν να εγκαταλείψουν τη χώρα τους και θα ήθελαν να εγκατασταθούν σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε στον Καναδά, στη Βραζιλία, στη Χιλή, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από εδώ λείπει βεβαίως η Ευρώπη. Η Σουηδική Προεδρία είπε ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των επανεγκατεστημένων ε, προσφύγων στην Ευρώπη. Η Επιτροπή αναθεώρησε επίσης τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων για να έχει μια πιο ε, ισχυρή πολιτική επανεγκατάστασης. Εγώ, όπως ε, ξέρετε, παρουσιάζω δύο εκθέσεις εξ ονόματος της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών για να διορθωθεί για να διορθώσουμε μάλλον τις πολιτικές χρειάζονται ε, μια σειρά μέτρων. Δύο βασικές αλλαγές είναι περιεχομένου, άλλες δύο διαδικαστικές. Η πρώτη είναι οι περιφερειακές προτεραιότητες. Μέσα στο πλαίσιο των, των περιφερειακών προτεραιοτήτων υπάρχουν και ανθρωπιστικές προτεραιότητες. Τις διατηρούμε αλλά στις προτεραιότητες αυτές δίνουμε μεγαλύτερη αυτονομία. Η Ευρώπη πρέπει να έχει μια στρατηγική παρέμβαση για την επανεγκατάσταση, βασικό χαρακτηριστικό και της εξωτερικής μας πολιτικής που επιτρέπουν την παρέμβαση σε κάποιες περιοχές ε, του κόσμου, ανοίγοντας τις πόρτες σε πολίτες κάποιων χωρών ή ανοίγοντας τις σχέσεις μας με κάποιες περιφέρειες δίνοντας τα κράτη-μέλη την δυνατότητα να θεσπίσουν ανθρωπιστικές προτεραιότητες. Ε, για παράδειγμα, ε, θύματα ε, βασανιστήριων, γυναίκες ή παιδιά, θύματα σεξουαλικής βίας, άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας. Δεύτερον, η διαβάθμιση. Υπάρχουν 10 κράτη-μέλη που ασκούν πολιτική επανεγκατάσταση στην Ευρώπη. Θα, θα θέλαμε και τα 27 να ακολουθήσουν μια πολιτική επανεγκαταστάσεως. Για το λόγο αυτό ζητούμε την αύξηση του αριθμού των προσφύγων ανακράτος μέλος για το πρώτο έτος, μια δεύτερη χρονιά με κάποια μικρή μείωση και μια τρίτη χρονιά με ισότιμη αντιμετώπιση όλων των κρατών ώστε αυτό το ενισχυμένο ποσό, να, η αύξηση του ποσού δηλαδή, να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη βιωσίμων προγραμμάτων επανεγκατάστασης. Τώρα, οι διαδικαστικές αλλαγές. Η Επιτροπή μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία κατεπήγοντος για την επανεγκατάσταση προσφύγων όταν υπάρχει μια ανθρωπιστική καταστροφή ή μια ανθρωπιστική κρίση. Μέχρι τώρα η διαδικασία ήταν ετήσια και ξέρετε ε, οι κρίσει δεν περιμένουν ε, το τέλος του χρόνου. Και το δεύτερο είναι το βασικό ζήτημα των κατεξουσιαδότης συμπράξεων. Εγώ να σας πω κύριε Επίτροπε ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να προχωρήσει πολύ γρήγορα τα θέματα κατεπήγοντος. Έχουμε πολύ ταχεία δυνατότητα αντι, ε, απάντησης, αντίδρασης στις προτάσεις κατεξουσιοδότησης πράξεων. Η Επιτροπή Εξωτερικών και η Επιτροπή Δημοσίων Ελευθεριών μπορεί να έχουν διαφορές ως προς τις, τις περιοχές προτεραιότητες. Αυτό μπορούμε να το ξεπεράσουμε, αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε να έρχεται η Επιτροπή και να μας λέει ότι η κατεξουσιοδότηση πράξης δεν πρέπει να καταγράφονται μεταξύ αυτών των σημαντικών πράξεων εξωτερικής πολιτικής ή δημοσιονομικής πολιτικής διότι θεωρείται ότι είναι πολύ γραφειοκρατική διαδικασία. Εμείς λέμε όχι. Πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό είναι τμήμα των κατεξουσιοδότηση πράξεων και κατά συνέπεια η Επιτροπή θα έπρεπε να προασπίσει την καταχώρησή τους και να μην δημιουργεί διαδικαστικού χαρακτήρα προβλήματα. Δεν θέλουμε το ζήτημα, τα ζητήματα αυτά να εμποδίσουν το να πετύχουμε τον κοινό μας στόχο, την αύξηση του αριθμού των προσφύγων που επανεγκαθίστανται. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ταβάρες. Οι επόμενοι ομιλητές, ο κύριος Μπούσουτιλ για δύο λεπτά έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Αυτό το πρόγραμμα εγκατάστασης που δημιουργείται καλύπτει ένα κενό που υπάρχει Χρειαζόμαστε το πρόγραμμα αυτό και πρέπει να σας πω πως με εκπλήσει το ότι το πρόγραμμα αυτό δεν υπήρχε μέχρι τώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν χώρε που μπορεί να μα δώσουν ένα καλό παράδειγμα. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, για παράδειγμα, έχουν ένα πολύ καλό πρόγραμμα επανεγκατάσταση, έχουν μακρά εμπειρία, μπορούμε να μάθουμε πολλά από αυτού. Τα προγράμματα αυτά, προφανώ, είναι πολύ σημαντικά. Διότι δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να δείξει το ανθρωπιστικό της πρόσωπο στον κόσμο. Υπάρχει κι άλλο σημαντικός λόγος ωστόσο. Ταυτόχρονα μειώνουμε την πίεση της, στις παράνο, των παράνομων ροών μετανάστευσης. Καλύπτουμε τις περιπτώσεις ανθρώπων που χρειάζονται προστασία και έρχονται σε εμά. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό το πρόγραμμα κατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να πάρουμε ανθρώπους από τη Λιβύα που αναζητούν μια διεθνή προστασία, ε, μειώνοντας κατά συνέπεια τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι αυτοί θα περάσουν τη Μεσόγειο παράνομα, διακινδυνεύοντας τη ζωή τους. Τους βοηθάμε λοιπόν τους ίδιους, βοηθάμε ταυτόχρονα και τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή τη στιγμή υφίστανται το δυσανάλογο βάρος της υποδοχής τους. Προφανώς το πρόβλημα αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί, να αντιμετωπιστεί με ένα άλλο πρόγραμμα, να συνοδεύεται μάλλον με ένα άλλο πρόγραμμα που θα βοηθήσει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αντιμετωπίζουν ένα δυσανάλογα μεγάλο ε, βάρος στην υποδοχή ετούντων άσυλων και προσφύγων επιτρέποντας την μεταφορά ανθρώπων που έχουν διεθνή προστασία σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή τη στιγμή υπάρχει και τρέχει ένα πιλωτικό πρόγραμμα για τη Μάλτα. Θα θεωρούσε ωστόσο ότι αυτό το έργο θα μπορούσε να ε, το μιμηθούν και άλλες χώρες της Ένωσης που έχουν παρόμοιες, παρόμοια προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έντσιο για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Ως... σε ευχαριστώ πολύ. Όσον αφορά το πέρασμα από το ΣΥΣ 1 στο ΣΥΣ 2 και σαν σκιώτης εισηγητής, θα ήθελα να συγχαρώ τον ε, εισηγητή, τον κύριο Κοέλιο, για το πνεύμα συνεργασίας που έδειξε και την εξαιρετική συνεργασία που είχαμε. Ευχαριστώ ιδιαίτερα και την Επίτροπο, την κυρία Μέλστρομ, καθότι από τότε που ανέλαβε τη θέση αυτή υπάρχει πολύ περισσότερη διαφάνεια και πνεύμα συνεργασίας. Η έλλειψη διαφάνειας και οι τρομερές καθυστερήσεις έχουν ε, πάρα πολύ καθυστερήσει την πρόεδρο των εργασιών μας. Η Επιτροπή δεν μπόρεσε να μας δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία όσον αφορά τη μεταφορά των δεδομένων. Δεν ξέρουμε επίσης αν οι δοκιμές που έγιναν ήταν επιτυχείς ή όχι. Υπάρχει λοιπόν μεγάλη αβεβαιότητα όσον αφορά την βιωσιμότητα αυτού του προγράμματος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την αρμοδιότητα να ελέγξει τον τρόπο δαπάνης των κοινοτικών κονδυλίων. Ζητήσαμε λοιπόν τα κονδύλια αυτά για το ΣΥΣ2 να μπουν στο αποθεματικό. Είναι θέμα ασφάλεια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να εκφράζει την άποψή του όσον αφορά την, πρόεδρο, την πρόοδο συγγνώμη, του ΣΥΣ2. Δεν είναι δυνατόν να αποτύχει το σχέδιο αυτό καθότι δεν υπάρχει αρκετή πολιτική βούληση ή διαφάνεια. Θα πρέπει να γίνει μελέτη μελέτη ωφέλειας και να μας δοθεί μια ημερομηνία για τις επόμενες φάσεις. Ευχαριστώ πολύ. κυρία Σντάνοκα, ένα, ένα μισή λεπτό. Για το SIS θα μιλήσω κι εγώ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, καταρχάς να ευχαριστήσω τον κύριο Κοέλιο για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η ομάδα μου εξ αρχής ήταν ε, εξαιρετικά επιφυλακτική ως προς την αποδοχή του SIS-2 λόγω των πολλών προβλημάτων στον τομέα της προστασίας των δεδομένων. Από ό,τι φαίνεται οι δοκιμές δεν έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν καθυστερήσεις, αύξηση του κόστους χωρίς θετικά αποτελέσματα. Ούτε καν υπάρχει συνένεση μεταξύ των ε, επιδογμόνων για την αξιολόγηση των δοκιμών. Η Γαλλία και η Γερμανία θεωρούν ότι δεν είναι επιτυχής. Κατά την άποψή μας η προσέγγιση του εισηγητού είναι σωστή, απολύτως σωστή. Πρέπει να είμαστε ε, ειλικρινείς, να δεχθούμε ότι οι δοκιμές και το έργο μπορεί να αποτύχει και να εξετάσουμε εναλλακτικέ λύσεις. Επίσης, να εξετάσουμε προσεκτικά γιατί απέτυχαν απέτυχε το σύστημα. Αν πρέπει να επενδύσουμε 30 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, το Κοινοβούλιο θα έπρεπε πριν από το αποφασίσει να έχει όλες τις ε, πληροφορίες που είναι αναγκαίες. Επίσης, πρέπει να υπάρξει μια ρήτρα λήξη. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να επενδύουμε σε διαβίου, σε συνεχιζόμενα προγράμματα. Πρέπει να υπάρχουν σαφή κριτήρια αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και ταχεία αντίδραση αν διαπιτωθεί ότι κάτι πάει λάθος ξανά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ένς για 1,5 λεπτό έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ. Καταρχήν θεωρώ και φυσικά αναφέρομαι στο θέμα SIS, ότι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και γεγονότα. Γνωρίζοντας το τι συμβαίνει με τις δοκιμές οι οποίες έχουν ξεκινήσει και τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών. Σε αυτό θα πρέπει να βασιστούμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποβάλει μία σειρά μέτρων και μέχρι τώρα διαπιστώσαμε ότι για τεχνικούς ή νομικούς λόγους τα κράτη-μέλη δεν μπορούν να ανταποκριθούν στους στόχους αυτούς. Και εδώ μιλώ εξ ονόματος της ε, γερμανικής ε, θέσης. Έτσι όπως έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή στην ε, Γερμανία, θεωρούμε ότι τα ποσά που έχουν δαπανηθεί είναι υπερβολικά. Δεν θέλουμε να υπάρξει αναβολή, περαιτέρω αναβολή μέχρι το 2013. Θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε ένα εναλλακτικό σύστημα η ομάδα των αριστερών έχει ήδη υποβάλει μία σειρά επιφυλάξεων και επικρίσεων όσον αφορά τον απόρριτο χαρακτήρα αυτών των στοιχείων, όσον αφορά τις μυστικές υπηρεσίες, τις υπηρεσίες πληροφοριών και την ανάμιξη των αρμοδιοτήτων που κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε με αυτήν την νέα πρόταση τα βιομετρικά στοιχεία, στοιχεία τα οποία κατά την άποψή μας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με τελείως διαφορετικό τρόπο αυτό που προτείνεται. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μέσερ Σμιτ είναι ο επόμενος ομιλητής, αλλά δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Ο επόμενος είναι ο κύριος Διαπολίνο, ο οποίος έβαλε τα ακουστικά του. Με ακούσατε, για δύο λεπτά έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Κυρία Επίτροπε, ο καθορισμός συνεπών προσεγγίσεων για να, έχουμε, για να δείξουμε μία ε, πραγματική αλληλεγγύη προς τα κράτη-μέλη αποτελεί μια βασική πρόοδο στην κοινωτική πολιτική για τη μετανάστευση. Ταυτόχρονα είναι ε, το ξεκίνημα μιας ευρύτερης διαδικασίας για την διεθνή προστασία των προσφύγων. Αν η διαδικασία αυτή αποβεί χρήσιμο με, το, με την εμπλοκή και της κοινωνίας των πολιτών θα εξαντληθεί από την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστηρίξη Ασύλου. Θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει ένας κατάλογος προτεραιοτήτων και στόχων με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μέτρα και κίνητρα και με επαρκή χρηματοδότηση για να μπορέσουν περισσότερα κράτη-μέλη από τα σημερινά δέκα να προσχωρήσουν στο πρόγραμμα επανεγκατάστασης χωρίς να ξεχνάμε την ανάγκη υγειονομικής προστασίας που θα περιλαμβάνει και κοινωνική κοινωνική προστασία υπερατόμων που συχνά υφίστανται ε, εξαιρετικά τροτές συνθήκες ζωής. Ταυτόχρονα θα μπορέσει να ε, επιτρέψει την ε, εξασφάλιση μιας οικογενειακής επανένωσης στη διαδικασία ένταξης. διαδικασία αυτή θα, στη διαδικασία αυτή είναι αναγκαία η συνεργασία μεταξύ των μερών για να υπάρξει ταχύτητα και ευελιξία στις διαδικασίες. Θέλουμε μια πιο δίκαια, πιο ρεαλίστρια και πιο αλληλέγγυα Ευρώπη που λαμβάνει υπόψη τις προσπάθειες των κρατών της νότιας κυρίως Ευρώπης ε, και τις προσπάθειες των κρατών μελών, των, κρατών, των τρίτων κρατών. Ταυτόχρονα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενισχύσει την προσπάθεια ε, σύναψη συμφωνιών συνεργασίας όπως έκανε πρόσφατα η Ιταλία με την Λιβύη και με άλλες χώρες. Δεν θεωρούμε ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος ε, για να περάσουμε από την ε, αλληλεγγύη που είναι συχνά μόνο θεωρητική στην πραγματική ουσιαστική διαχείριση από κοινού των μεταναστευτικών οδών. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κυρία Μπένεβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον συνάδελφο, τον κύριο Τάβαρες. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι λυπάμαι πάρα πολύ που τα κράτη-μέλη παρέχουν πάρα πολύ περιορισμένα μέτρα για την εγκατάσταση των προσφύγων. Υπάρχει πάρα πολύ ελλειπής υποστήριξη, πάρα πολύ ελλειπής συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών με αποτέλεσμα να αυξάνεται και το κόστος της επιμέρους αντιμετώπισης του φαινομένου. Η πολιτική αυτή φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί με ολοκληρωμένο τρόπο στην Ευρώπη. Εμείς θα πρέπει σαν Ευρωπαίοι να προτείνουμε ένα νέο ελκυστικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που να διακατέχεται από το πνεύμα της αλληλεγγύης πρόγραμμα σε σχέση με τη χρηματοδότηση, τη εγκατάσταση και όλες αυτέ οι δραστηριότητε θα πρέπει να συντονίζονται με έναν κεντρικό τρόπο. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριος τα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους οι οποίοι εργάζονται σκληρά με αυτήν την ιστορία η οποία δεν σταματάει ποτέ και τον κύριο Κοέλιο και τους υπόλοιπους καθυστερήσεις οι οποίες μας ανησυχούν. Τι άλλο θα μπορούσε να χαρακτηρίσει καλύτερα τις διαχειριστικές ικανότητες του κυρίου Μπαρόζο στην Επιτροπή από αυτήν την κατάσταση. Πιστεύω θα πρέπει να μάθουμε από την κατάσταση αυτή και να δούμε τι προτείνει εδώ με μια δημιουργία μιας νέας υπηρεσίας στο Τάλιν με τον προγραμματισμό που θα γίνεται από εκεί όσον αφορά τις ε, υπηρεσίες πληροφορικής. Η ολοκλήρωση στον τομέα αυτό σίγουρα θα προτείνει την προστασία των δεδομένων αλλά και μια ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του φαινομένου. Η κυρία Μάλστρομ, η οποία έχει αναλάβει το θέμα αυτό, ελπίζω να είναι σε θέση, τουλάχιστον έτσι πιστεύω, να το ολοκληρώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Δίας Δεμέρα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα σας τα πω τηλεγραφικά. Πρώτον, να συγχαρώ τον κύριο Κοέλιο. Η διαδικασία έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί πριν τις 39 του. Πρέπει να αλλάξουν πριν λήξει η προθεσμία τα εργαλεία. Δεύτερον, καμία πρόταση της Επιτροπής δεν θέτει προθεσμία και δεν κατ και δεν καταργεί τις ρήτρε πάυσης ε, της αρχικής, ε, του αρχικού κειμένου. Τρίτον, πρέπει να υπάρξει μία προθεσμία για την μετάβαση που να διευρυνθεί ενδεχομένω αν χρειαστεί μέσω επιτροπολογία. Τέσσερα, η διαδικασία δεν ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι πολύ κακό. Πέμπτον, αγνοούνται τα αποτελέσματα των τεστ για το SIS2. Το Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερωθεί για αυτά. Έκτον, Υποστηρίζω για τους λόγους αυτούς την πρόταση του εισηγητή και την προειδοποίηση για το ενδεχόμενο παρέμβαση του ελεγκτικού συνεδρίου αν αποτύχει το έγγραφο. Για την έκθεση Ταβάρε τώρα, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων και την Επανεγκατάσταση. Και πάλι να συγχαρώ τον κύριο Ταβάρε. Βασικό πρόβλημα, η έλλειψη εσωτερικής ελληνικής στην Ένωση. Πρέπει να προχωρήσουμε προσεκτικά σε ό,τι αφορά τις ενισχύσει σε κράτη-μέλη που υποδέχονται για πρώτη φορά πρόσφυγες, ιδίως ε, εξετάζοντας τις ε, συγκριτικές, τους συγκριτικούς μισούς. Τα μέτρα αυτά που, του κύριου Ταβάρες που υποστηρίζω καταρχήν απαιτούν καταρχάς μια προκαταρκτική και μελετημένη ε, οικονομική εξέταση. Η κυρία Κιγιόμ, 1,5 λεπτό. Αγαπητοί συνάδελφοι, Νομίζω ότι θα είμαστε υπέρ της επαναδιάρθρωσης ε, των Ευρωπαϊκών Ταμείων υπέρ των προσφύγων. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να συγχαρώ τον Κάρλος Κοέλο και τον Αλβάρες για το έργο που έκαναν. Η ψηφοφορία επί του σχεδίου αυτού υπογραμμίζει την ανάγκη των χωρών μελών να καταβάλουν κάθε προσπάθεια ώστε να καλύψουν ένα διπλό κενό ε, τόσο από πλευρά των χωρών μελών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όσο και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακριβώς ε, ε, θα πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες ώστε να αντιμετωπιστούν οι τραγικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν οι ε, πρόσφυγες στις χώρες ε, αυτές. Έτσι λοιπόν ε, είμαστε υπέρ της προσπάθειας αυτής με τη δέσμευση ότι όλες οι χώρες μέλη θα αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί ε, όπως λέει η κυρία Μάλστρομ. Βεβαίως η πρόκληση είναι δύσκολη δεδομένου ότι οι χώρες μέλη διαθέτουν ελάχιστα ε, μέσα. Ωστόσο βασιζόμαστε στη δική σας αποφασιστικότητα και δέσμευση. Η εσωμάτωση των προσφύγων είναι κλειδί για την ε, ε, υλοποίηση και την επιτυχία αυτού του προγράμματος το οποίο πρέπει να γίνει υπό τις καλύτερες συνθήκες και οι χώρες μέλη θα πρέπει να επιδείξουν μεγάλη ε, δέσμευση δεδομένου ότι ε, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να ανασχέσουμε αυτήν την μαζική ροή προς την Ευρώπη. Ευχαριστώ. Τελευταίος ο κύριος Όμπεν Μάγκερ. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ όσον αφορά τη χώρα μου την Αυστρία πιστεύω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε όλες αυτές τις προτάσεις για την επανεκατάσταση των προσφύγων ιδιαίτερα για χώρες οι οποίες βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως παραδείγματος χάρη χώρες που δέχονται πρόσφυγες από τις ανατολικές χώρες, από την Ουκρανία κτλ. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο αυτό με απόγνωση ή με αδιαφορία. Σήμερα γνωρίζουμε ότι υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες πολιτικές οι οποίες είναι διαφορετικές από τη μία χώρα στην άλλη. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι διαρκώς θα συνεχίζουν να έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πρόσφυγες, καθότι το βιωτικό μας επίπεδο και οι οικονομικές συνθήκες είναι ελκυστικές. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι προστασία των εξωτερικών συνόρων. Αυτό είναι προϋπόθεση. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Τελείωσε η κοινή συζήτηση και θα ξεκινήσει η διαδικασία Catch the Eye. Κάποιοι ομιλητές έχουν ζητήσει το λόγο. Έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μας και οι ομιλητές είναι ο κύριος Λούχαν. Για να δω. Πρόεδρε, συνάδελφοι, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων στηρίζεται στη συνεργασία και αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. Τούτο ωστόσο δεν μπορεί να γίνει αναχώρα μόνο. Απαιτείται μια ευρωπαϊκή κοινή πρωτοβουλία. Γι' αυτό για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται το πρόγραμμα επανεγκατάστασης. Χρειαζόμαστε ένα αποτελεσματικό και ουσιαστικά αλληλέγγυο πρόγραμμα, ούτως ώστε να υπάρχει ένα πλαίσιο που θα δείχνει ότι τα κράτη-μέλη θα εμπλακούν πραγματικά στην επανεγκατάσταση προσφύγων. Η προσπάθεια των κρατών μελών για την εισδοχή, για την ε, ένταξη προσφύγων θα πρέπει να συνοδεύεται και από οικονομικά κίνητρα. Με τα μέτρα αυτά θα δείξουμε πραγματική αλληλεγγύη της Ένωσης για το παγκόσμιο πρόβλημα των προσφύγων και να ενθαρρύνουμε την συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξεπερνάτε το χρόνο ομιλία που είναι ένα λεπτό για τη διαδικασία Eye. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο κύριος Μαρινέσκο. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα κι εγώ να κάνω μια παρατήρηση καταρχήν, η οποία αφορά τον συνάδελφο που κάθεται εδώ αριστερά. Και πιστεύω ότι το ίδιο μπορεί κανείς να πει και όσον αφορά έναν Ιρλανδό, ο οποίος διαπράττει ένα δίκημα και ο οποίος θα πρέπει να σταλεί στην χώρα από την οποία προέρχεται. Έχω την εντύπωση ότι αυτό όμως δεν μπορεί να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2011. Η ερώτησή μου λοιπόν προς την Επιτροπή είναι ποιες είναι οι συνέπειες όσον αφορά την προσχώρηση χωρών που ακόμα δεν είναι μέλη του Σέγγεν δεν ανήκουν στο χώρο Σέγγεν. Σήμερα δεν μπορεί η Επιτροπή να μας δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία όσον αφορά το ξεκίνημα λειτουργίας του συστήματος SIS-2. Επιπλέον δαπάνες, επιπλέον επενδύσεις φαίνεται να είναι απαραίτητες. Και αν καταφέρουμε να χρησιμοποιήσουμε το SIS-1 συν το SIS-2, θα πρέπει να υπάρξει καλύτερο συντονισμός διαχείρισης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Μέσερ Σμιτ. Σας ευχαριστώ. Πριν από ένα χρόνο ήμασταν όλοι μαζί στην προεκλογική εκστρατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βεβαίως το θέμα του Σέγγεν έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προεκλογική αυτή εκστρατεία καθότι οι ψηφοφόροι της Ευρώπης είναι εξαιρετικά δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση τους εσωτερικούς ελέγχους, τον έλλειπτο έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα που είναι ελλειπής καθώς και τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζει ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα πρέπει να προσχωρήσουν στο Σέγγεν. Βεβαίως ξέρω ότι πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη, αλλά προς ποιον πρέπει να επιδείξουμε αυτήν την αλληλεγγύη, γιατί εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη εκμετάλλευση του συστήματος, του συστήματος το οποίο οργανώσαμε Βεβαίως να δείξουμε αλληλεγγύη, να δείξουμε αλληλεγγύη προς αυτούς που απειλεί σήμερα η Επιτροπή. Η κυρία Αντζελίλη έχει το λόγο, λέει Πρόεδρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το να έχει η Ευρώπη μια κοινή πολιτική ασύλου και μια στρατηγική επανεγκατάσταση σημαίνει να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματα του ανθρώπου και ταυτόχρονα να περιορίσουμε την παράνομη μετανάστευση. Χάρη λοιπόν, ε, ευχαριστώ στους, ε, τους εισηγητές και την Επίτροπο Μάρστρομ. Τώρα πλέον έχουμε ένα εξαιρετικό εργαλείο για τις χώρες δύο ε, εκείνες που βρίσκονται στη λεκάνη της Μεσογείου, την Ιταλία για παράδειγμα, που μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να έχουν ούτε μια πραγματική ελεγγύη από τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, ούτε μια δίκαιη κατανομή των ευθυνών. Πρέπει να υποστηρίξουμε τις πολιτικές αυτές με επαρκή προπολογισμό και με σοβαρούς ελέγχους των υλοποιήσιμων των προγραμμάτων που υλοποιούνται και με ουσιαστικές ε, δράσεις. Για τα ανθρώπινα δικαιώματα να κλείσω πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες ομάδες. Παιδιά, ανηλίκους, θύματα ε, εμπορίας, θύματα ε, ακροτισμένου γεννητικών οργάνων, κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι εξετάζει η κυρία Μάλστρομ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βέλτσερ έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, πιστεύω πραγματικά ότι τα μέσα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν αρκούν. Μιλάμε για 30 εκατομμύρια, τα οποία θα πρέπει να διατεθούν για την αντιμετώπιση όλων των θεμάτων που αφορούν την μετανάστευση και τους πρόσφυγες. Το θέμα είναι τα εξωτερικά σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διάτρητα χιλιάδες πρόσφυγες από τρίτες χώρες μπαίνουν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς κανέναν έλεγχο. Θα ήθελα λοιπόν πραγματικά να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή οικογένεια και τα επιχειρήματα ότι χρειαζόμαστε μετανάστες και πρόσφυγες είναι κάτι το οποίο σήμερα δεν μπορούμε να το υποστηρίξουμε. Αν ανοίξουμε τις πόρτες καταλαβαίνετε ότι το φαινόμενο αυτό είναι κάτι που δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε οι οικονομικοί μετανάστες. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι που πλημμυρίζουν την Ευρώπη. Και πραγματικά το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν είναι ένα πολύ μικρό τμήμα αυτών των δαπανών. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Μην ξεπερνάτε σας παρακαλώ πολύ το χρόνο ομιλία σας, γιατί ο χρόνος που διαθέτουμε είναι ελάχιστος. Ο κύριος Πάσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το σύστημα πληροφοριών του Σέγγεν για το οποίο θα μιλήσω είναι το εξής. Το σύστημα αυτό λειτουργεί εδώ και χρόνια. Μας κόστισε ε, πολλά. Καθίσταται όλο και πιο ακριβό και δεν γνωρίζουμε και τα αποτελέσματα. Είναι λοιπόν καιρός να γίνει ένας έλεγχος για να δούμε αν το σύστημα αυτό είναι ικανό να λειτουργήσει αποτελεσματικά. Αν είναι χρήσιμο για την Ευρώπη και μετά να εξετάσουμε τι, βήματα, τι περαιτέρω βήματα θα λάβουμε. Χρειάζεται δηλαδή να ελέγξουμε καταρχήν, διότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η παράνομη ε, μετανάστευση ε, όπως ε, έτσι ώστε νόμιμα να εγκαθίστανται οι πραγματικά έχοντες ανάγκη και ετούντες άσυλο. Τούτο τούτο λεχθέντος ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στις ε, νέες χώρες μέλη. Ε, ευχαριστώ πολύ. Το θέμα αυτό συνδέεται άμεσα με θέματα ασφαλείας. Συζήτησα προηγουμένως για την έκθεση Μάλκε, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα όσον αφορά τις επιπλέον θέσεις για την γραμματεία και την ετήσια αύξηση των θέσεων του προσωπικού καθώς και κάποιες επιπλέον αποδοχές. 1.500 ευρώ το μήνα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θα πρέπει να επιβαρύνουν το φορολογόμενο. Μιλάω για την έκθεση Μάλκη και προηγουμένως το συμφώνησα αυτό με το προσωπικό του Προεδρείου. Όχι, το είπα ήδη κύριε Συνάδελφε, δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε. Ο κύριο Μπόρις είναι ο τελευταίο ομιλητή για τη διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΗ και έχετε το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ του τους δύο εισηγητές. Και θέλω να πω το εξής. Σήμερα δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το σύστημα ΣΥΣ. Το σύστημα ΣΥΣ 2 θα πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή. Γι' αυτό λοιπόν εμείς υποστηρίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο νέος κώδικας για τις θεωρήσεις περιλαμβάνει και βιομετρικά στοιχεία. Έτσι το ΣΥΣ 2 θα επιτρέπει την ε, γρήγορη και ε, το γρήγορο και αποτελεσματικό έλεγχο των στοιχείων των ελεγχομένων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πολύ πρόσφατα υιοθετήσαμε μέτρα, μέτρα τα οποία ε, επιτρέπουν ε, επιτρέπουν την επικοινωνία και την σύνδεση για την ανταλλαγή πληροφοριών στο χώρο Σέγγεν. Ελπίζω λοιπόν ότι η Κομισιόν θα λειτουργήσει ανάλογα. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η συζήτηση και δίνω τώρα το Ευχαριστώ όλα τα μέλη για την υποστήριξη και τα σχόλια πάνω στα δύο διαφορετικά μένα αλλά πολύ σημαντικά θέματα. Αρχίζω με το ΣΥΣ 2. Είμαι η πρώτη που θα αναγνωρίσω ότι ε, πράγματι είναι ένα τεράστιο θέμα, πολύ σύνθετο, πολύ δύσκολο. Ίσως τα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα στο παρελθόν, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή είμαστε δεσμευμένοι να δουλέψουμε με έναν πολύ διαφανή, και, ε, διαφανή τρόπο. Και ακριβώς η Κομισιόν το έθεσε αυτό με αυτόν τον τρόπο στο Συμβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξε στα συμπεράσματα ε, ότι η δοκιμή η πρώτη δοκιμή ήταν επιτυχής. Αυτή τη στιγμή οι εμπειρογνώμονες καλούνται να αποτιμήσουν και να καθορίσουν τις προϋποθέσεις για τις χώρες μέλη και να καθοριστούν πιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για να προχωρήσουμε. Και η πρόταση θα γίνει στις 3 και 4 Υπουργείου προς τους Υπουργούς, οι οποίοι θα το συζητήσουν και θα υπάρξει περαιτέρω αξιολόγηση τούτου μετά το καλοκαίρι. Και όλες αυτές και καθ' όλο αυτό το διάστημα θα υπάρξει διαφανής επικοινωνία με το Κοινοβούλιο και τους συζητητές. Ε, η ε, αξιολόγηση για Βουλγαρία και Ρουμανία θα γίνει με βάση το ΣΥΣΑ 1 και εντωμεταξύ ενημερώνονται οι χώρες αυτές από αυτού. Επίσης προετοιμαζόμαστε και ελπίζουμε ε, να υπάρξει πετυχημένη δοκιμή δύο το φθινόπωρο. Οι επαφές μας είναι ανοιχτές και έχουμε τα αυτιά και τα μάτια ανοιχτά για να ε, στεφθεί με επιτυχία. Εν τω μεταξύ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλα τα μέλη για την υποστήριξή τους, να ευχαριστήσω τον κύριο Κουέλο και σας διαβεβαιώ για μία ακόμα φορά για τη δέσμευσή μας να λειτουργήσουμε με απόλυτη διαφάνεια και σε συνεργασία με, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την μετεγκατάσταση, ε, εκπλήσωμε που αναφέρθηκε από κάποιο μέλος ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε με ενιαίο τρόπο το θέμα των προσφύγων. Ε, αυτή τη φορά απλώς κάνουμε την προσπάθεια να έχουμε έναν πιο συντονισμένο τρόπο και να κάνουμε πιο ευφυή χρήση των κονδυλίων σε συντονισμό με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ώστε πραγματικά να αλλάξουν τα πράγματα για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται ή παγιδεύονται σε πάρα πολύ δυσχερείς καταστάσεις. Ε, μόλις ε, πέρσι 747.000 άτομα βρέθηκαν σε αυτήν την κατάσταση. Είναι τεράστιες οι ανάγκες όπως είπε ο κ. Φλάτρα. Νομίζω ότι συμφωνούμε πάνω στην, στο νόημα και το σκοπό αυτού του Ταμείου και πιστεύω ότι η πρόταση μπορεί να υιοθετηθεί χωρίς καθυστέρηση. Αρκετοί βουλευτές αναφέρθηκαν στην εσωτερική αλληλεγγύη, η οποία είναι αλληλένδετη βεβαίως, αλλά είναι διαφορετικό θέμα. Αναγνωρίζω την ανάγκη τούτου. Επίσης, η Κομισιόν έχει κάνει ήδη προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση και έχουμε προτείνει την προσωρινή διακοπή του κανονισμού του Δουβλίνου. Έχουμε θεσπίσει το Ευρωπαϊκό Γραφείο Υποστήριξης με έδρα τη Μάλτα. Αργότερα φέτος έχουμε ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο αξιολογούμε και συμφωνώ ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους να λειτουργήσουμε σε πιο μόνιμη βάση, σε συνεργασία με τις χώρες μέλη. Πάντως η Κομισιόν θα το εξετάσει και θα εξετάσουμε επίσης ε, έναν γενικότερο εσωτερικό μηχανισμό αλληλεγγύης ε, για του χρόνου. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το πρόγραμμα της μεταγκατάστασης. Ευχαριστώ πάντως τον κύριο Κουέλο και τον κύριο Ταβάρης, όπως επίσης και τον κύριο Άλβαρες, για το έργο τους σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό θέμα και ελπίζω ότι θα ολοκληρώσουμε το ταχύτερο δυνατό. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Τώρα οι εισηγητές. Καταρχάς ο κύριος Κουέλιο. Δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα ευγενικά τους λόγια. Κύριε Επίτροπε, το Κοινοβούλιο γνωρίζει ότι κληρονομήσατε το θέμα αυτό. Έχουμε εμπιστοσύνη και στην ικανότητα και στην εξυπνάδα σας για να το ολοκληρώσετε. Εκτιμούμε επίσης την προσπάθεια διαφάνειας ε, που καταβάλλετε, την οποία προσπάθεια υπογράμμισαν ε, πολλοί συνάδελφοι νωρίτερα. Σε ό,τι αφορά την προθεσμία, αυτό είναι ένα κακό μήνυμα. Αν τα νέα εργαλεία δεν έχουν προθεσμία, η μόνιμη και εσαή παράταση των προθεσμιών από την Επιτροπή δεν έχει νόημα. Πρέπει να τηρηθούν οι προθεσμίες. Μια προθεσμία που μπορεί να θέσει το Κοινοβούλιο. Να θέσουμε την προθεσμία εάν για κάποιο λόγο αυτή η προθεσμία δεν μπορέσει να τηρηθεί, να επανέλθετε ζητώντα παράταση. Αλλά το να δίνουμε παρατάσει έτσι η Κίκαιο έτυχε χωρί προθεσμία αποτελεί κατά την άποψή μου πολύ κακό μήνυμα για όλου. Η ιδέα σα να υπάρχει ε, να μην είναι μια συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνολικού Προγράμματος ε, είναι ενδιαφέρουσα. Ωστόσο, να σας πω ότι η πρόταση του Κοινοβουλίου ήταν συνέπεια μιας μετάβασης που ήταν χειρότερη από την αρχική πρόταση της Επιτροπής. Η αρχική πρόταση, παρότι περιόριζε την σύνθεση της Επιτροπής, επέτρεπε να, μετέχουν, ε, να μετέχει το Διοικητικό Συμβούλιο του Προγράμματος σε Άλλε δραστηριότητε. Εάν οι αρμοδιότητε του οργάνου αυτού περιοριστούν, θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε μόνο υπό βασικές προποθέσει και εγγύησει. Ευχαριστώ. Ο κύριο Τάβαρες. Ευχαριστώ και εγώ, κυρία Πρόεδρε, και ευχαριστώ όλους όσοι μίλησαν, την Επίτροπο. Νομίζω ότι αν, εφόσον υπάρξει βούληση για την, το, ο λόγος για τον οποίο υπάρχει βούληση για την επανεγκατάσταση προσφύγων είναι διότι η, η συζήτηση για τη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι δύσκολη και βλέπουμε ότι μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα αυτό και για μας και για τους πρόσφυγες. Όσοι έχουν πάει σε στρατόπεδα προσφύγων και έχουν δει τα παιδιά που ζουν εκεί χρόνια και χρόνια, χάνοντας χρονιέ σπουδών που θα μπορούσαν να έχουν στην Ευρώπη, δείχνει πόσο επίγωσα είναι η συζήτηση. Ελπίζω επίσης να λυθούν τα διαδικαστικά ζητήματα. Βάσει της συνθήκη. Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι αρκετό. Απαιτείται μία γραμμή προπολογισμού, όχι μόνο για το πρόγραμμα επανεγκατάστασης προσφύγων Αυτά προσπαθήσαμε να αντιμετωπίσουμε ε, στην έκθεση πρωτοβουλία που είχαμε υποβάλει. Η ποιότητα. Η ποιότητα στην ένταξη των προσφύγων είναι πολύ ε, σημαντική και απαιτεί συνεργασία με τις ΜΚΟ, την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, απαιτεί δε επίλυση των γραφειοκρατικών προβλημάτων συντονισμού. Το γεγονός ότι τα παιδιά που βρίσκονται στο στα στρατόπεδα προσφύγων δεν πηγαίνουν στο σχολείο και το γεγονός ότι καθυστερούμε ε, οφείλεται στο ότι τα κράτη-μέλη διστάζουν γιατί χρειάζονται πολύ χρόνο για να ε, ε, συμφωνήσουν στην επικύρωση των ταξιδιωτικών εγγράφων των προσφύγων. Αυτό μπορεί να γίνει ωστόσο μέσω ε, μια ειδική αρμοδιότητα στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξη Ασύλου που θα δημιουργήσει μια μονάδα επανεγκατάσταση με κάποιου λίγου υπαλλήλου και που θα επιτρέπει να ολοκληρώνουν τι διαδικασίε επανεγκατάσταση, να παρουσιάζει τι βέλτιστε πρακτικέ και να εμπλέκει τα κράτη-μέλη στη διαδικασία αυτή, συντονίζοντά τη με την Υπηρεσία Εξωτερικών Αρμοδιοτήτων, με την Διπλωματική Υπηρεσία τη Ένωση για να διευκολύνει διευκολυνθεί η επανεγκατάσταση. Όταν αποφασίσουμε και εφόσον αποφασίσουμε την επανεγκατάσταση δεν μπορούμε να την καθυστερούμε λόγω διοικητικών ή γραφειοκρατικών καθυστερήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο περατώσαμε και την κοινή συζήτηση. Στις 12 θα λάβει χώρα η ψηφοφορία. Και τώρα περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η έκθεση του συναδέλφου Άλβες. Πρόκειται για την θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού προγράμματος και τα μέτρα για την γεωργία στις εξόχως απόκεντρες